Okay, colleagues, uh, please. Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε σας παρακαλώ πολύ για να ξεκινήσει η συνεδρίασή μας. Καλωσορίσατε μετά τις θερινές διακοπές. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω πάλι όλους. Αγαπητοί συνάδελφοι, ας ξεκινήσουμε όμως τώρα τη συνεδρίασή μας. Θα ήθελα να κάνω μια σειρά από ανακοινώσεις. Μια σειρά λοιπόν από ανακοινώσεις όσον αφορά τη σημερινή ημερήσια διάταξη. Ευχαριστώ Τόμας. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θα κάνω μια σειρά ανακοινώσεων όσον αφορά τη σημερινή μερίσια διάταξη και συνέχεια θα κάνω μία-δύο ανακοινώσει ε, όσον αφορά την μεταναστευτική προσφυγική κρίση προκειμένου να δούμε λίγο τι συμβαίνει και να έχουμε και τη δυνατότητα να κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις. Θα κάνω και κάποιες ακόμα επίσημες ανακοινήσεις στη συνέχεια τη μερίσια διάταξη. Καταρχάς, Κάποιε αλλαγές για την ημερήσια διάταξη, οι οποίε πρέπει να εγκρίνεται σήμερα το πρωί. Έχουμε ένα νέο σημείο 4.1. Τριμερής διάλογος όσον αφορά ορισμένες πτυχέ του τεκμηρίου αθότητα και του δικαιώματο παράσταση του κατηγορωμένου στη δίκη του. Στις 9 και 20 θα εξετάσουμε το ζήτημα αυτό. Έχουμε ήδη καθυστερήσει λίγο. Σημείο 6 τη ημερήσια διάταξη η ψηφοφορία για την κινητοποίηση του μέσου ευελιξία για τα προσωρινά μέτρα στον τομέα τη διεθνού προστασία υπέρ τη Ιταλία και τη Ελλάδα είναι σημείο το οποίο αναβάλλεται όσον αφορά την ασφαλή χρήση των συστημάτων τηλεχειριζόμενων αεροσκαφών, το σημείο 7 δηλαδή, θα το ψηφίσουμε πριν από το σημείο 5 και τα σημεία 11 και 12 της της διάταξης ενημέρωση από την εκτελεστικό διευθυντή της Frontex είναι σημεία τα οποία αναβάλλονται δεν είναι διαθέσιμος ο διευθυντής της Frontex, είναι στην Ελλάδα αυτές τις μέρες για προφανείς λόγους. Θα προσπαθήσει να έρθει σε κάποια επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μας και θα έχει δυνατότητα να μας ενημερώσει για την κατάσταση. Αγαπητοί συνάδελφοι, επίσης, να αναφέρω τώρα ορισμένα πράγματα όσον αφορά την ε, κρίση την οποία αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή και ξέρω ότι ορισμένοι συνάδελφοι θέλουν να πάρουν το λόγο. Την επόμενη Τετάρτη έχουμε την δήλωση για την κατάσταση της Ένωσης από τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα μας απασχολήσει προφανώς το ζήτημα αυτό πάρα πολύ, αλλά η διάσκεψη των Πρόεδρων ήδη σήμερα θα αποφασίσει αν θα προβλεφθεί μια επιπλέον συζήτηση την επόμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια για την προσφυγική κρίση. Μέχρι τις 12 λοιπόν σήμερα θα γνωρίζουμε. Επίσης, όσον αφορά ιδιαίτερα τη δική μας την ε, Επιτροπή, οι συντονιστές θα αποφασίσουν ε, τη Δευτέρα στη συνεδρίασή τους τι επιπλέον στοιχεία θέλουν ε, να δούνε όσον αφορά την ανταπόκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κρίση, όσον αφορά την ανταπόκριση σε όλα αυτά τα ζητήματα που έχουν προκύψει. Η συνεδρίαση λοιπόν αυτή των συντονιστών θα λάβει χώρα τη Δευτέρα. Να επενθυμίσω τώρα στους συναδέλφους ότι θα συνεδριάσουμε στις 14 του μηνός, μάλλον στις 14 Σεπτεμβρίου έχουμε το Συμβούλιο των Υπουργών Εσωτερικών και Δικαιοσύνης για τη μεταναστευτική κρίση και θα πρέπει να δούμε και εμείς πώς θα προετοιμαστούμε για αυτή τη συνεδρίαση και θα ψηφίσουμε την επόμενη εβδομάδα μια έκθεση όσον αφορά το ζήτημα κατανομής των προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να έχουμε τον απαραίτητο χρόνο και ακόμα και τη δυνατότητα να κάνουμε μια επιπλέον συνεδρίαση της Επιτροπής μας προκειμένου, αν κρυθεί δυνατό, να συζητήσουμε εκ νέου το μηχανισμό ανακατανομής των προσφύγων που προβλέπει να συζητήσει η της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 14 Σεπτεμβρίου. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να κινηθούμε πολύ προσεκτικά, πολύ μεθοδικά, δεν θα πρέπει να συγχαίουμε τα ζητήματα μεταξύ τους και θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ήδη ενώπιον μας έχουμε μια πολύ σημαντική έκθεση Όσον αφορά την μετανάστευση, ήδη θα πρέπει να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε την έκθεση αυτή στις δύο δυνατότητες που θα έχουμε να την εξετάσουμε 15 και 23 Σεπτεμβρίου. Εγώ θα συναντήσω κατά πάση πιθανότητα την επόμενη εβδομάδα τον αρμόδιο επίτροπο και θα μπορέσουμε το ζήτημα αυτό να το συμπεριλάβουμε και στην ε, συνάντηση της 14 Σεπτεμβρίου. Ήθελα να αναφερθώ στα σημεία αυτά γιατί γνωρίζω το, το ζήτημα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρω ότι υπάρχουν μεμονωμένοι συνάδελφοι που είτε μόνοι τους είτε στα πλαίσια της πολιτικής τους ομάδας είτε σε εθνικό επίπεδο ασχολούνται ενεργά με το ζήτημα αυτό και θεώρησα θα έπρεπε να πω αυτά τα εισαγωγικά λόγια. Δεν ξέρω αν τώρα θέλει κάποιος να πάρει το λόγο για να προσθέσει επιπλέον σημεία στην ημερήσια διάταξη, να κάνει παρατηρήσεις στην ημερήσια διάταξη προτού αυτή εγκριθεί. Κορνίλια παρακαλώ. Ήθελα να πω κάτι για τα προβλήματα των προσφύγων, αλλά μπορώ να το κάνω και μετά. Μετά τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Πώς το προτιμάτε, τι είναι σωστότερο. Μου είναι αδιάφορο, μπορώ και άμεσα να το πω. Αμέσως. Να το κάνω λοιπόν. Um, Αν θέλετε τώρα να το αναφέρετε, γιατί θα θέλαμε μετά να συζητήσουμε. Για τα θέματα προσφύγων, έτσι. Ωραία, συνεχίστε λοιπόν τώρα. Λοιπόν, συμβαίνει το εξή. Είναι πολύ καλό βρίσκω ότι εμείς ευθύς εξ αρχής ε, συμφωνούμε για μια διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί. Δεν είναι η χρονική στιγμή όπου ο ένας πρέπει να κατηγορεί τον άλλον από πλευράς κρατών μελών. Αυτό δεν οδηγεί πουθενά. Θα έπρεπε αυτή την κλιμακωμένη κατάσταση, την ένταση σε σχέση με τα προβλήματα των προσφύγων πολύ νυφάλια και ήρεμα να τα συζητήσουμε. Αυτό πρέπει να καταφέρουμε. Οι εικόνες που το καλοκαίρι είχαν διαβιβαστεί σε όλα τα κράτη-μέλη και σε εμά στη Γερμανία που σπίτια όπου θα βρίσκαν καταφύγιο πρόσφυγες είχαν ε, πέσει θύματα εμπρισμού και είχαν καεί και τώρα, τώρα στην αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων στη Γερμανία μπορούμε να ολοκληρώσουμε αυτά και για κάθε κράτος μέλος να δούμε τι πρέπει να γίνει πώς να το πω, δεν μπορούμε με προκατηλημένες απόψεις ε, και ιδεολειψίες να προχωρήσουμε. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια σοβαρή αντικειμενική συζήτηση. Πρέπει να συζητήσουμε για τις ε, σημασιολογικές αυτές έννοιες και τις προσεγγίσεις ε, όσον αφορά αυτά τα ζητήματα. Υπάρχουν θέματα που άμεσα πρέπει να δράσουμε για την ανθρωπιστική ανάγκη που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Παιδιά κυρίως, παιδιά που βρίσκονται σε μια καταστροφική ολέθρια κατάσταση όσον αφορά τους πρόσφυγες. Και πρέπει να τους χορηγηθεί υποστήριξη, συνδρομή και βοήθεια. Τώρα για την επόμενη εβδομάδα key debate, περαιτέρω συζήτηση, υποστηρίζουμε την πρόταση του Προέδρου μας της Κοινοβουλευτικής μας Επιτροπής. Εμείς ως συντονιστές, αυτή είναι η παράκλησή μου, θα ήθελα τη Δευτέρα να τοποθετηθούμε με δικές μας προτάσεις επ' αυτών. Τι δηλαδή τους επόμενους μήνες θα κάνουμε και πώς θα συμφωνήσουμε να προχωρήσουμε. Θέλουμε τα εξή θέματα να συμφωνήσουμε ώστε να τεθούν υπό εξέταση. Ανάλυση της συνολικής κατάστασης των προσφύγων συμπεριλαμβανομένη τη άμεση βοήθεια και των άμεσων μέτρων τη Ευρωπαϊκή Ένωση και χρηματοοικονομικών μέτρων που πρέπει να συζητηθούν για να βελτιωθεί η κατάσταση στα κράτη-μέλη. Δεύτερον, συζήτηση για την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Ακόμα και καγκελάριο τη Γερμανία, κυρία Μέρκελ, είπε ότι το σύστημα αυτό είναι προβληματικό όσον αφορά ποσοστώσεις ε, και μετεγκαταστάσεις ε, και πρέπει να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Αυτές τις τροπολογίες θα τις καταθέσουμε ως προτάσεις τη Δευτέρα. Οι συντονιστές ε, των άλλων ομάδων και αυτοί να συμμετάσχουν ώστε να έχουμε ένα πίνακα να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Um, Ευχαριστούμε Κορνίλια, δεν ξέρω αν και άλλοι συνάδελφοι θέλουν να πάρουν το λόγο ή ενδεχομένως τη Δευτέρα να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους στην Συνεδρία των ιστών, γιατί ήδη σε 9.30 θα πρέπει να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Σε ευχαριστούμε, Κορνίλια, και θα προτιμάσουμε τη συνεδρίαση αυτή για τη Δευτέρα. Ανακοινώσεις τώρα του Πρόεδρου. Να εγκρίνουμε λίγο τις συστάσεις των συντονιστών σύμφωνα με το άρθρο 205. Οι ακόλουθες εκθέσεις έχουν δοθεί στον Χουάν Φερνάντο Λόπες Αγουιλάρα ενωσιακό κώδικα για τις κατά πολέμηση της απάτης κατά των χρηματοοικονομικών συμφερόντων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυρία Σίλβια Ιβόν Κάουφμαν θα είναι η συγγήτρια όσον αφορά τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την, τον ομοιόμορφο μορφότυπο για τις θεωρήσεις. Και τέλος η κυρία Τερίσα Χιμένες Μπεχερίλ Μπάριο από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θα είναι η συγγήτρια για, την, για το σχέδιο εφαρμοστικής απόφασης του Συμβουλίου δεν πρόκειται καν να προσπαθήσω να διαβάσω όλες αυτές τις χημικές ενώσεις. Πρόκειται πάντως για ένα σύστημα νέων μέτρων ελέγχου για συγκεκριμένες χημικές ουσίες. Νομίζω ότι είναι ο μεγαλύτερος, ο πιο μακροσκελής τίτλος έκθεση που έχω δει ποτέ. Ο κύριος Μάικλ Μπόνι από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θα είναι εισηγητής πάλι για μία έκθεση η οποία φέρει ένα πολύ μεγάλο τίτλο και επίσης θα είναι εισηγητής ε, για μία νέα έκθεση όσον αφορά μέτρα ελέγχου και η κυρία Ιντβέλτ θα είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία ενός νέου μηχανισμού για την παρακολούθηση της εφαρμογής των θεμελωρίων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου. Ο κύριος Άνβερτ από τους ε, Πρασίνους θα είναι υπεύθυνο προ τη σύσταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, όσον αφορά την συμφωνία ΤΙΣΑ για τι υπηρεσίε και ο Μάκλ Μόνι από το ΕΛΚ θα είναι εισηγητής για τη γνωμοδότηση όσον αφορά την ψηφιακή ενωσιακή αγορά και ο κύριος Βόητα από τους μη εγγεγραμμένους θα είναι εισηγητής για τη γνωμοδότηση όσον αφορά την ε, ε, πάρκια προστασία των καταναλωτών για το νέο ψηφιακό περιβάλλον. Μπορούμε να εγκρίνουμε αυτές τις συντάσεις των ιστών, θεωρώ πως ναι, επομένως εγκρίνονται. Όσον αφορά το χρόνο ψηφοφορίας, προτείνω να κινηθούμε ηλεκτρονικά, να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά, επομένω σας έχετε μαζί στις κάρτες σας. Πρωτού όμως προχωρήσουμε στην ψηφοφορία, θα ήθελα να ακούσουμε μία ενημέρωση όσον αφορά τους ανεξελίξει τριμερείς διαλόγους και να ξεκινήσω από την εισηγήτριά μας Κατερίνα Κινίτσι όσον αφορά την παρουσίαση της πρόοδου των τριμερών διαπραγματεύσεων για τις δικονομικές εγγύσεις για τα παιδιά που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών. Στις 14 Ιουλίου Λεβεχώρα, χώρα ο τελευταίος τριμερής διάλογος. Δεν ξέρω αν Κατερίνα μπορείς εν συντομία να μας ενημερώσεις. Ευχαριστώ Κλοντ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Στις 14 Ιουλίου όντως είχαμε την τέταρτη συνεδρίαση του τριμερού ε, διαλόγου, τη της διαπραγματεύση υπό υπολήξιμβοριανής προεδρία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Προεδρία αυτή γιατί δείχνει ένα πολύ θετικό πνεύμα συνεργασία μέχρι στιγμή και από ό,τι φαίνεται έχει αναλάβει μια σημαντικότατη δέσμευση για το ζήτημα αυτό. Προσπαθεί δηλαδή να βρει λύσει λαμβάνοντα υπόψη την θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να καταφέρουμε να καταλήξουμε σε ένα οριστικό κείμενο το συντομότερο δυνατό γιατί ουσιαστικά ελπίζουμε αυτή τη στιγμή να καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε το κείμενο αυτό κατά πάσα πιθανότητα κατά τη διάρκεια του φθινοπόρου ή τουλάχιστον κατά τη διάρκεια του, της Προεδρίας ε, του Λουξεμβούργου. Συμμετείχαν ε, λοιπόν ε, όλοι στον τριμερή αυτό διάλογο. Έγινε μια πολύ σημαντική προπαρασκευαστική εργασία στα πλαίσια των τεχνικών επαφών που είχαμε και μου δόθηκαν και κάποιες συγκεκριμένε ενδείξεις από τους σκιώδεις συγγητές και τους ευχαριστώ για την συμβολή τους. Δεν θα ήθελα να μπω τώρα σε τεχνικές λεπτομέρειες, να σας πω απλώς ότι καταφέραμε να συμφωνήσουμε ήδη για ορισμένα σημεία με το Συμβούλιο, θεμελιώδη θεωρώ σημεία όσον αφορά τις δικονομικές εγγύσεις των ύποπτων ή κατηγορούμενων παιδιών. Ένα πολύ σημαντικό σημείο είναι ότι πλέον έχουμε έναν ορισμό όσον αφορά το τεκμήριο της ε, ανηλικότητας, της, ε, της ηλικίας ουσιαστικά του παιδιού ή του ανήλικα. Ένα άλλο σημαντικό σημείο που το οποίο καταφέραμε να πετύχουμε συμφωνία είναι το δικαίωμα ενημέρωσης και πληροφόρησης. Έγινε μια ενδελεχή συζήτηση για το ζήτημα αυτό, αλλά καταφέραμε τελικά να καταλήξουμε σε μια συμφωνία και είπαμε ότι ο ύποπτο ή κατηγορούμενος ανήλικος θα πρέπει να λαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες χωρίς βέβαια να κατακλείζεται από πάρα πολλές περιττές πληροφορίες, αλλά με τις πληροφορίες εκείνες που έχουν να κάνουν πραγματικά με τα δικονομικά του δικαιώματα κατά τη διάρκεια της ποινική διαδικασίας. Ένα άλλο σημαντικό σημείο είναι η ατομική αξιολόγηση του ανήλικα, Πάλι εδώ πέρα αναφερθήκαμε σε συγκεκριμένους στόχους και στο περιεχόμενο της αξιολόγησης αυτής και ξέρετε ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η ατομική αξιολόγηση γιατί προβλέπει τελικά τη δυνατότητα να βρεθούν συγκεκριμένα μέτρα για τον συγκεκριμένο ανήλικα που θεωρείται ύποπτος ή κατηγορούμενος. Συμφωνεί επίσης ε, επετεύχθη όσον αφορά και τις ιατρικές εξετάσεις. Έγινε πάλι μία σε βάθος συζήτηση. Από ό,τι φάνηκε υπήρχαν ορισμένες χώρες στο Συμβούλιο οι οποίες αντιστέκονταν πάρα πολύ στην πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ήθελε ουσιαστικά να διευρύνει περισσότερο το δικαίωμα αυτό της ιατρικής εξέτασης. Δεν προβλέπεται πλέον αυτή η γενικότερη αναφορά στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, το medical care, αλλά παρόλα αυτά καταλήξαμε σε ένα θετικό συμβιβασμό. Σε κάθε περίπτωση δηλαδή υπογραμμίζεται η αρχή ότι ο ανήλικος ή το παιδί που έχει στερηθεί την προσωπική του ελευθερία έχει δικαίωμα σε πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Επομένως, θεωρούμε ότι και αυτό αποτελεί ένα πολύ θετικό συμβιβασμό. Προσπαθούμε επίσης αυτή τη στιγμή να καθορίσουμε περισσότερο πώς θα διαπραγματευτούμε συγκεκριμένα άρθρα τα οποία παραμένουν ακόμα ανοιχτά, για παράδειγμα, η εξειδικευμένη κατάρτιση όλων των δικαστικών και όλων εκείνων οι οποίοι εργάζονται στα πλαίσια της ποινική διαδικασίας κάθε φορά που εμπλέκονται παιδιά. Εκκρεμούν βέβαια δύο σημεία αρκετά αμφιλεγόμενα, το δικαίωμα δικαστικής συνδρομής μέσω δικηγόρου, καθώς επίσης και το ίδιο το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας αυτής ε, όσον αφορά την ε, τυπολογία των ε, εγκλημάτων που εκδικάζονται και όσον αφορά την τελική έκβαση της δικαστικής διαδικασίας. Θα συνεχιστούν επί των δύο αυτών σημείων οι συζητήσεις και πιστεύω ότι με τη βοήθεια της Προεδρίας του Λουξεμβούργου θα καταφέρουμε να πετύχουμε και για τα δύο αυτά σημεία συμβιβασμό και κατά αυτόν τον τρόπο θα οριστικοποιήσουμε, θα ολοκληρώσουμε το κείμενο. Και προφανώς είμαι στη διάθεση των συναδέλφων για περαιτέρω διευκρινήσεις. Ευχαριστώ. Λόγω χρόνου αν δεν σας πειράζει, θα πάμε κατευθείαν στο επόμενο για τις, ε, η κατάσταση της, ε, ε, των, της παραμονής ανθρώπων που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών. Η Ευχαριστώ Πρόεδρε, καλημέρα σε όλους. Είναι καλό που επιστρέψαμε, ελπίζω να ήταν καλό το καλοκαίρι, ειδικά για σας κύριε Πρόεδρε, γιατί αυτό το φθινόπωρο θα είναι πολύ δύσκολο για όλους μας. Ε, βλέπω λοιπόν ε, ε, ότι μάλλον είναι καλό να είμαστε όλοι ευδιάθετοι. Στις 16 Ιουλίου είχαμε τον τέταρτο ε, τριημερή διάλογο για το θέμα των επιστημόνων, ε, ερευνητών δηλαδή και φοιτητών από ε, τρίτες χώρες. Έγινε σε καλό πνεύμα, μέσα σε πνεύμα συνεργασίας και τα τρία θεσμικά όργανα δεσμεύτηκαν για την οριστικοποίηση του θέματος αυτού μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Εφόσον όλοι λοιπόν είμαστε πεπισμένοι ότι αυτός ο φάκελος, αυτό το θέμα θα είναι ε, προς όφελος κάθε κράτους μέλους ε, και θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε και πάλι η συζήτηση για το πεδίο εφαρμογή της οδηγίας και αποφασίστηκε ότι θα υπάρξει περαιτέρω διαπραγμάτευση στον επόμενο τριμερή διάλογο γιατί το θέμα αυτό είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο. Επίσης καταφέραμε να συμφωνήσουμε σε θέματα που έχουν να κάνουν με την αίτηση για θεώρηση, την ε, παρουσίαση των εγγράφων στην επίσημη γλώσσα, την ε, διαδικασία προέγκρισης, τις επαρκή, τους επαρκείς πόρους για τα άτομα που καταθέτουν αίτηση, τον ορισμό των ε, μελών της οικογένειας και τη διαφάνεια. Πολύ καλά λοιπόν πήγαν τα πράγματα εκεί. Τώρα όσον αφορά τους λόγους απόρριψης ή μη ανανέωσης, ε, είχαμε κάποια πρόοδο αλλά παραμένουν κάποια εκκρεμή ζητήματα. Ε, μεταξύ αυτών, ε, το, ο, λόγος ε, που έχει προσθέσει το Συμβούλιο στο άρθρο 18F που λέει ότι αν υπάρχουν επαρχικές λόγοι να θεωρείται ότι παραμένει στο χώρο, στον τόπο κάποιος για λόγους ε, σοβαρούς, ε, μπορεί να παραμείνει. Αυτό βέβαια ε, παρα... βγαίνει εκτός του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας και δεν μπορούμε απλώς να το αποδεχτούμε. Επίσης, Χρειάζονται και άλλες συζητήσεις για τη διεύθυνση στην χώρα φιλοξενίας, για την αγορά εργασίας και την εργασία των φοιτητών. Μετά τον τριμερή διάλογο ε, πήγα στην ε, ανεπίσημη συνεδρίαση της ΚΕΦΑ στο Λουξεμβουργό, όπου εκεί είχαμε διμερείς συναντήσεις με εκπροσώπους από διαφορετικά κράτη-μέλη. Νομίζω ότι έγιναν ε, οχτώ τέτοιες συναντήσεις με μέλη των κυβερνήσεων των κρατών μελών και πραγματικά ήταν μια καλή ευκαιρία για να μπορέσουμε να μιλήσουμε με τα κράτη-μέλη που ήταν εκεί. Και για μένα προσωπικά για να βελτιώσω την αγάπη μου για το Λουξεμβούργο και ειδικότερα για το Σέγγεν. Έτσι λοιπόν ήταν μια καλή άσκηση. Ο επόμενος τριμερής διάλογος θα γίνει στις 29 Σεπτεμβρίου κύριε Πρόεδρε. Αδειμονώ λοιπόν και αδειμονώ ε, για, να μπορέσω για τη συνεργασία που θα έχουμε φέτος το φθινόπωρο με τους Σκιώδης. Ως τώρα είχαμε πολύ καλή συνεργασία, θεωρώ λοιπόν ότι μπορούμε να συνεχίσουμε μέχρι τέλους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Σεσίλια, συνάδελφοι, τουλάχιστον ένας έχει ζητήσει το λόγο, όμως ε, όπως έγινε και με την προηγούμενη έκθεση δεν θέλω να κάνουμε τις ερωτήσεις τώρα γιατί η ψηφοφορία είναι στις 9.30. Έχουμε Επίσης, άλλη μια έκθεση για τριμερή διάλογο που δεν είναι στην ημερήσια διάταξη, όμως πρέπει να την ακούσουμε ε, από τη Λατνή Κρίσπερκ, η οποία είναι συγκήτρια για την ε, οδηγία για το τεκμήριο της αθωότητας. Παρακαλώ να έχουμε μια ενημέρωση και για αυτό το τριμερή διάλογο, αν είναι δυνατόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Μετά από αυτές ε, τις δύσκολες διακοπές όπως είπαμε, όπως λέμε στη Γαλλία, Έχουμε αυτή την ε, ε, παρουσίαση της οδηγίας για το τεκμήριο αθωότητας. Το Νοέμβρη του 2013 θυμάστε ότι η Κομισιόν δημοσίευσε το νομοθετικό πακέτο για, τα για το δικονομικό δίκαιο που μεταξύ άλλων περιείχε και αυτή την οδηγία. Το 2014 το Δεκέμβρη ε, υιοθετήθηκε η γενική προσέγγιση για αυτή την οδηγία και το Μάρτιο του 2015 η Επιτροπή μας ενέκρινε με μεγάλη πλειοψηφία τη θέση της ε, για αυτό το κείμενο. Ξεκίνησε άμεσα ο τριμερής διάλογος και υπήρξε και μια πολύ καλή έτσι, ατμόσφαιρα συνεργασίας ε, στις διαπραγματεύσεις μεταξύ μας για να προχωρήσουμε σε αυτό το κείμενο κλειδί για την ε, σεβασμό ε, της άμυνας στην Ευρώπη και για το, ε, και τον Απρίλιο και τον Μάρτιο, Μάιο υπό τη Λετωνική Προεδρία είχαμε άλλους δύο τριμερείς διαλόγους, τους ευχαριστώ. Στον πρώτο τριμερή διάλογο εξετάσαμε χωρίς να κάνουμε ανταλλαχή και λεπτομερή εξέταση του άρθρου 14 της οδηγίας. Μετά το Μάιο πήγαμε και εξετάσαμε τα άρθρα 1 έως 5 και ε, προχωρήσαμε. Είχαμε κάποια ε, συμφωνία, κυρίως για το άρθρο 3, ειδικότερα για το πεδίο εφαρμογής, ε, το άρθρο 2, αλλά παραμένει ακόμα σε κάποια σημεία ανάγκη εξέτασης. Μετά, στο άρθρο 5 και άλλη, φορά, και άλλη μια φορά, ε, πάλι για το προσωπικό και υλικό κομμάτι του πεδίου εφαρμογή της ε, οδηγίας, πάλι άρθρο 2, η παρουσίαση επίσης των υπόπτων ε, ενώπιον κάποιες δικαιοδοσίας, αυτό είναι το άρθρο 4. Ο τρίτος ε, διάλογος ξεκίνησε την πρώτη μέρα της Λουξεμβουργικής Προεδρίας, την 1η Ιουλίου και εξετάσαμε τα υπόλοιπα άρθρα Φυσικά έγινε κάποια πρόοδος ε, στα άρθρα 6 και 7, όμως οι διαπραγματεύσεις ε, παραμένουν ε, δύσκολες, ειδικότερα για το δικαίωμα διατήρησης της σιωπής άρθρο 6, τη μία αποδοχή τεκμηρίων όταν γίνεται αυτή η απόκτηση με παραβίαση του δικαίου της Επίσης, η η κρίση δίμην, Επίσης η παρουσία και η γρήγορη και αποτελεσματική εφαρμογή, ε, ε, η γρήγορη ε, αποτελεσματική δράση των σκιωδών. Υπάρχουν λοιπόν κάποια πολύ σημαντικά στοιχεία, κυρίως για το πεδίο εφαρμογής, το δικαίωμα σιωπής και την δίκαιη ρήμεν. Επίσης για τη μία αποδοχή των τεκμηρίων, ε, ζητώ συγγνώμη που είμαι τόσο τεχνική πρωί-πρωί, αλλά είμαι στη διάθεσή σας για να συζητήσουμε ε, σχετικά με, το, με τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς είναι οι εκθέσεις ε, και σας ευχαριστούμε πολύ για την ανάλυση. Ωραία. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που άκουσαν όλες αυτές τις ε, εκθέσεις, τις αναφορές για τους τριμερείς διαλόγους. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη σκληρή δουλειά που έχετε κάνει και ευχαριστούμε και για τις εκθέσεις. Υπάρχει κάποιο θόρυβο, αλλά μάλλον επειδή πρόκειται να ε, επίκειται μια ψηφοφορία αυτή τη στιγμή. Αγαπητοί συνάδελφοι, αν θέλετε να ησυχάσετε λιγάκι, να καθίσετε. Να σας εξηγήσω και πάλι ότι η ψηφοφορία θα είναι ηλεκτρονική και γι' αυτό θα πρέπει να έχετε τις κάρτες σας. Όποιος δεν έχει την κάρτα του να μου το πει παρακαλώ. Όλοι την έχουν, ωραία. Οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε, να σταματήσουμε για ένα, για λιγάκι μάλλον. Okay, colleagues, if you're ready, we can... Συνάδελφοι, αν είστε έτοιμοι μπορούμε να προχωρήσουμε για την ε, πρώτη ψηφοφορία είναι η ασφαλής χρήση των συστημάτων ελεγχειριζόμενων αεροσκαφών και για τα μη επανδρομένα αεροσκάφη είναι μια έκθεση μη... Ε, ιδίας πρωτοβουλίας. Είστε όλοι έτοιμοι? Το μικρόφωνο σας είναι ανοιχτό. Είστε έτοιμοι? Όλοι έτοιμοι λοιπόν. όσοι είναι όρθιοι και τριγυρίζουν γύρω-γύρω και δεν, ε, ή δεν παίρνουν μέρος στην ψηφοφορία, παρακαλώ να καθίσετε. Δεν είστε ακόμη όλοι στις θέσεις σας. Παρακαλώ μπορείτε να καθίσετε για την ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Περνάμε στην ψηφοφορία. Συμβασμός 5. Είναι όλα ηλεκτρονικά. Ανοίγει η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Περιμένω την κάρτα μου, οπότε ε, θέλω να ε, συνταχθώ με τα υπόλοιπα μέλη των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών με ανάταση της χειρός. Θα την έχω σε ένα δευτερόλεπτο την κάρτα μου. Κάποιος άλλος που θέλει να πει κάτι. Μια πιο ήσυχη ανακοίνωση ακούω. <laughs> Αλλαγή μικροφόνο. Μάλλον πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή. Να ξεκινήσουμε και πάλι. Λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία. Περιμένω μέχρι να είναι όλοι έτοιμοι. Να ξεκινήσω και πάλι να ρωτά, ρωτώντας αν όλοι έχετε την ηλεκτρονική σας κάρτα και είστε έτοιμοι για την ψηφοφορία. Καλημέρα, Φρανκ. Hm. You have to ask again. Yeah, yeah. Okay, we're going to open the boat. Άρχεται η ψηφοφορία σε λιγάκι, λοιπόν. Από ό,τι είδα, δεν ψήφισαν όλοι. Όσοι έχετε ηλεκτρονική κάρτα, παρακαλώ να είστε εδώ, να είστε στην αίθουσα και να είστε και ξύπνοι, παρακαλώ. Συμβιβασμό 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Ξεκινάμε από την αρχή. πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβιβασμό 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Ζητώ συγγνώμη. Πρώτα η τροπολογία 23. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραστε της Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 6. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 7. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα στις ψηφοφορίες. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8, άρχεται η ψηφοφορία. Ε, συμβαστική τροπολογία 8, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 9, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 10. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 11. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 12. Άρχεται η ψηφοφορία. πέρα της ψηφοφορία εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 13. Άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία τώρα. Πέρα της ψηφοφορία εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 14. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 15. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική ε, τροπολογία μάλλον 53. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 16. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα τη ψηφοφορία εγκρίνεται. Ε, η ιταλική σκέψη της συμβαστικής 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας τη ψηφοφορία. εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 2. Πρώτο μέρος. Χωριστή ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Δεύτερο μέρος συμβαστικής τροπολογίας 2. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 3 των αιτιολογικών σκέψεων άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Για την ε, τροπολογία 12 άρχεται η ψηφοφορία. Η 12. Πέρα της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 17 είναι προφορική ε, τροπολογία η λέξη νομιμότητα αντικαθίσταται από τη λέξη αναγκαιότητα, legitimacy necessity. Άρχεται η ψηφοφορία. Δεν υπάρχουν ε, αντιρρήσεις για αυτή την προφορική τροπολογία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Και η τελική ψηφοφορία για το συν... Α, συγγνώμη, πρώτα η τροπολογία 18. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Ζητώ συγγνώμη, πρέπει να ξανακάνουμε την τροπολογία 18. Τροπολογία 18. Άρχεται η ψηφοφορία και πάλι. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. για το τροποποιημένο κείμενο άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Και περνάμε αμέσως συνάδελφοι. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Περνάμε κατευθείαν στις τροπολογίες για τον προϋπολογισμό. Εισηγητής ο Πέτρον Νίδεμιλ. Ξεκινάμε με την τροπολογία 5916. Ψηφίζουμε. Ποιο είναι το πρόβλημα. Δεν υπάρχει. Τι είναι. Ωραία, ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Ψηφίζουμε. Προχωράμε. Τροπολογία 5916. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ποιο, τι πρόβλημα υπάρχει. Working amendment and the other one is Sorry, colleagues, I think you maybe have some Συνάδελφοι, ίσω υπάρχει κάποια σύγχυση. Ξεκινάμε με τι τροπολογίε για τον προπολογισμό, προπολογισμό τροπολογίες επί του προπολογισμού. Εντάξει, έχετε τη σωστή, τον σωστό πίνακα ψηφοφορία μπροστά σα. Λοιπόν, πρέπει να βρείτε τι τροπολογίε για τον προπολογισμό. Ξεκινάμε με την τροπολογία 5916. Εντάξει, Βρισκόμαστε όλοι στην ίδια σελίδα για να ξεκινήσουμε. Ωραία, πολύ καλά τώρα πια. Λοιπόν. Okay, let's open. Πολύ καλά, ας ξαναξεκινήσουμε. Έχετε όλοι το σωστό πίνακα ψηφοφορία στα χέρια σας. Εντάξει, είναι σημαντικές αυτές οι ψηφοφορίες. Δεν θέλω να βιαστούμε και να γίνουν κάποια λάθη. Λοιπόν, έχετε τις σωστές, ε, τους σωστούς πίνακες, ξεκινάμε πάλι. 59-16 τροπολογία. Άρχεται η ψηφοφορία. Λοιπόν, ξεκινάμε ξανά, έτσι. Okay, the vote is now closed. That is adopted. That is adopted. Um, the... Εγκρίθηκε η τροπολογία 59-18. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας Απορρίφθηκε αυτή. 59-46 τροπολογία άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα εγκρίθηκε. Τροπολογία 59-47 τώρα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίθηκε. Τροπολογία 59-19. Άρχεται. The vote Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 59-87. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. 59-91. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 59-86. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Περνάμε τώρα στην συμβαστική τροπολογία. Πάμε στην τροπολογία 59-72. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 59-38. Άρχεται. The Πέρας. That is rejected. Απορρίφθηκε. Και τώρα συμβιβαστική τροπολογία α άρχεται Πέρας ψηφοφορίας εγκρίθηκε ο συμβιβασμό. Τροπολογία 59, 22 τώρα. 59, 22. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας Αποτέλεσμα απορρίφθηκε. Τροπολογία 5983. Άρχεται η ψηφοφορία. 5983. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας απορρίφθηκε. Τώρα 59-82 άρχεται. Πέρας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 59-23 άρχεται. Πέρας. απορρίφθηκε. Τροπολογία 59-24. Άρχεται. Πέρας. Απορρίφθηκε. Περνάμε στο συμβιβασμό Β. Άρχεται η ψηφοφορία. Βρίσκεται ο συμβιβασμό Β. 59-70. Άρχεται η ψηφοφορία. 59-70. Άρχεται, παρακαλώ. Θα ήθελα να είναι σαφές για όλους επιτέλους ώστε να ψηφίσετε σωστά. Ψηφίζουμε την τροπολογία 5970, εντάξει. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε. Συνεχίστε η ψηφοφορία για να ικανοποιηθείτε όλοι. Εντάξει, πέρας ψηφοφορίας τώρα. Απορρίφθηκε η 5970. Πάμε στην τροπολογία 5979. Άρχεται. Τροπολογία 59-79. Πέρας ψηφοφορίας τώρα. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 59-40. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 59-45. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα απορρίφθηκε. 59-68 τροπολογία άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 59-88. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 59-89. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 59-26. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε τροφολογια 59 59-49. Άρχεται η ψηφοφορία. Ένας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Περνάμε στο συμβιβασμό γάμα. Σι. Άρχεται η ψηφοφορία παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 59-51. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 59-52. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. 59-53 τώρα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. 59-90. Άρχεται. Πέρας. απορρίφθηκε. 59 Το πρωί 5904 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας απορρίφθηκε. Τροπολογία 59, 54. Τροπολογία 59, 54. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία τώρα 59. 59-69. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε η τροπολογία αυτή. Τροπολογία 59-55. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 59-05. Άρχεται η ψηφοφορία. Σας ζητώ συγγνώμη συνάδελφοι, θα πρέπει να επαναλάβουμε την, πληφορία, την ψηφορία για την 5928. Έκανα λάθος πριν. 5928. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5929 αυτή ψηφοφορία. The vote is closed. Πέρας. That is rejected. Απορρίφθηκε. 59-42. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. 59-43. Άρχεται η ψηφοφορία. Είχαμε την τροπολογία 5943, εντάξει. Πέρας ψηφοφορίας τώρα. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 5944. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. 5956, 59-56. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. εγκρίθηκε. Περνάμε τώρα στην Ευχαριστώ για αυτή την συμμετοχή σας. Συνεχίζουμε. colleagues, we go straight to the draft opinion. Λοιπόν, πάμε στην έκθεση γνωμοδότησης. Πάλι συντάκτης ο Πέτερ Νίντεμιλ, τοπολογία 3. Άρχεται η ψηφοφορία επ' αυτής. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας απορρίφθηκε και αυτή. Τώρα η τροπολογία 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα εγκρίθηκε. Τροπολογία 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 7. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 8. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 6. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα απορρίφθηκε. Τροπολογία 9. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 10. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε τροπολογία 11. 11 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Ο συμβιβασμός Hey, α, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Συμβιβασμός α είπαμε. Ε, α. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Περνάμε στην παράγραφο 5. Στο εδάφιο 5, παράγραφος 5, όπως τοποποιήθηκε. άρχεται η ψηφοφορία επ' αυτού. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίθηκε, λέει ο πρόεδρος. Συγγνώμη διορθώνει ο πρόεδρος. Απορρίφθηκε, μάλιστα. Απορρίφθηκε λοιπόν. Πάμε τώρα στην παράγραφο 5, τροπολογία 16 και 17. Είναι ταυτόσιμες. Υπέρ αυτών λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκαν. Τροπολογία 19. η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 18. η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. απορρίφθηκε. Τροπολογία 20. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 21. Άρχεται. Πέρας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 22. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 23. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 24. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 25. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 26. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 27. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 28. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 29. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Και η τελική ψηφοφορία τώρα. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε στην τελική ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία. Συγχαρητήρια στον Πέτερ Νίντεμιρ για το έργο που επετέλεσε. Σας ευχαριστώ συνάδελφοι για τη συμμετοχή σας. Ολοκληρώνονται οι ψηφοφορίες. Ο Τόμας Ντουντόφσκι θα μας κάνει τώρα μια σύντομη ανακοίνωση. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί συνάδελφοι, σας ζητώ συγγνώμη το μόνο που ήθελα να πω είναι ότι ο να ευχαριστήσω τον Πίτερ Νίντερ Μούλερ για την καταπληκτική συνεργασία που είχαμε. Και είναι και τα γενέθλια του Πίτερ σήμερα, επομένω χρόνια του πολλά. Χρόνια σου πολλά για τα γενέθλιά σου, Πίτερ. Να το πω και στη γλώσσα σου. Thomas, that was very elegant. Thank you very much. Πολύ ευγενικό εκ μέρους σου. Ευχαριστούμε πολύ, Thomas. you never meet, but, but I propose again to, uh, to organize a leader working group after the... Colleagues, um, if we could... Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε τώρα σας παρακαλώ πολύ. Πρέπει να προχωρήσουμε με τα υπόλοιπα σημεία της ημερήσιας διάταξης. Πρέπει να καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε σήμερα το πρωί την ημερήσια διάταξή μας. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στα υπόλοιπα σημεία που έχουμε προς εξέταση, παρακαλώ πολύ καθίστε και οι υπόλοιπε συζητήσεις να συνεχιστούν εκτός εθούσης. Περνάμε τώρα στα σημεία 13 με 19 της ημερήσιας διάταξης. Αγαπητοί συνάδελφοι, για άλλη μια φορά σας παρακαλώ πολύ, σταματήστε όλες αυτές τις συζητήσεις. Τόμας, ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Αγαπητοί συνάδελφοι, ησυχάστε παρακαλώ πολύ. Περνάμε στα επόμενα σημεία της σημερινής διάταξης όσον αφορά το ζήτημα αμοιβαιότητας μορισμένες τρεις χώρες στον τομέα της πολιτικής θεωρήσεων. Έχουμε μια έκθεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπου γίνεται μια αξιολόγηση των διαφόρων συμφωνιών διευκόλυνσης χορήγησης θεωρήσεων, ιδίως όσον αφορά τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Αναφερόμαστε λοιπόν σε καθεστώτα διευκόλυνσης και απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης. Θα εξετάσουμε επίσης και την κατάσταση όσον αφορά τις θεωρήσεις για τη Γεωργία και την Ουκρανία και στο τέλος, αν ησυχάστε, θα καταφέρουμε να ενημερωθούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μάλλον δεν ενδιαφέρεται όμως κανείς από ό,τι βλέπω. Σας παρακαλώ πολύ καθίστε και θα ακούσουμε όπως σας έλεγα τέλος της παρατηρήσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις συμφωνίες διευκόλυνσης χορήγησης θεωρήσεων ή απαλλαγής από το καθεστώς θεωρήσεων για την Κολομβία και το Περού. Σας παρακαλώ πολύ, οι συζητήσεις που δεν έχουν σχέση με τη μίληση διάταξη να γίνονται εκτός εθούσης. Επίσης, θα πρέπει να ενημερωθούμε και εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για όλες τις διεθνείς συμφωνίες σχετικά με τις θεωρίες που συνάπτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και έχουμε μάλιστα και την πρόσφατη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κοινοβούλιο κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την κατάσταση του Μαυρικίου και την δυνατότητα μεταφοράς κάποιων ύποπτων πειρατών. Και για το ζήτημα αυτό είπε το δικαστήριο ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενημερώνεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Διαφορετικά οποιαδήποτε απόφαση δεν θεωρείται έγκυρη. Επαναλαμβάνω λοιπόν για άλλη μια φορά ότι δεν υπάρχει απλώς η δυνατότητα υποβολής αιτήματο ενημέρωση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά υπάρχει και η θεσπισμένη πλέον υποχρέωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο να μας ενημερώνουν για όλες αυτές τις διεθνείς συμφωνίες. Μπορούμε καταρχά λοιπόν να δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συνέχεια θα ακούσουμε και τα μέλη. Ο κύριο Νίλσεν νομίζω ότι είναι παρόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ή ο κύριο Πάλμεν. Και οι δύο, μάλιστα. Και οι δύο είναι παρόντε. Πολύ ωραία. Ποιο από του δύο θέλει να πάρει πρώτο το λόγο, παρακαλώ. Ο κύριο Πάλμεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι αναπληρωτή διευθυντή όσον αφορά το τμήμα θεωρήσεων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριο Νίλσεν, ο συναδελφό μου, είναι εδώ μαζί μου, ο οποίο είναι υπεύθυνο για κάποια άλλα ζητήματα. Εγώ θα σα μιλήσω κυρίω για το καθεστώ αμοιβαιότητα όσον αφορά τι θεωρήσει και για κάποιε άλλε διεθνεί συμφωνίε. Όσον αφορά το καθεστώ αμοιβαιότητα με ορισμένε τρίτε χώρε στον τομέα τη πολιτική θεωρήσεων, θα μπορέσω να σα πω κάποια πράγματα και στη συνέχεια θα αναφερθεί και ο συναδελφό μου στο ζήτημα απελευθέρωσης των θεωρήσεων. Όσον αφορά λοιπόν το ζήτημα της αμοιβαιότητας. Όπως ξέρετε, έχουμε έναν αθεωρισμένο μηχανισμό για την αμοιβαιότητα που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το Δεκέμβριο του 2013. Αυτός ο αθεωρημένος μηχανισμός έχει ως στόχο να δημιουργήσει ένα πιο πάγιο καθεστώς και μια δυνατότητα μεγαλύτερη και πιο γρήγορη αντίδραση τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε περιπτώσει μη αμοιβαιότητα. Δηλαδή κάθε έξι μήνες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει είτε να εγκρίνει μια εκτελεστική απόφαση, πράξη, όπου θα προβλέπεται αναστολή εξάμηνη του καθεστώτος μη υποχρέωσης θεώρησης, εφόσον υπάρχει απαλλαγή για το συγκεκριμένο ε, κράτος, τρίτο κράτος, και θα πρέπει να εξηγείται για ποιο λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε σε αυτή την πράξη ή για ποιο λόγο αποφάσισε ότι δεν έπρεπε να εγκρίνει τελικά μία εκτελεστική πράξη. Κάθε έξι μήνες λοιπόν υποβάλλονται εκθέσεις όσον αφορά τα μέτρα αυτά και αφού περάσουν 24 ε, ε, μήνες τότε πρέπει να ληφθεί μια οριστική απόφαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω πράξεις εξουσιοδότησης για την μόνιμη κατάργηση πλέον του καθεστώτος ε, μη υποχρέωσης θεώρησης. Ήδη από την Απρίλιο 2014 υπάρχει το καθεστώς αυτός, από τότε που άρχισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλαδή να κοινοποιεί γνωμοδοτήσεις όσον αφορά την μία αμοιβαιότητα σε σχέση με τρίτες χώρες. Εμείς έχουμε λάβει μέχρι στιγμής ειδοποιήσεις από τη Βουλγαρία, την Κροατία, την Κύπρο, την Πολωνία και τη Ρουμανία, πέντε δηλαδή κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιπτώσεις μία μηδεότητας θεωρήσεων σε σχέση με πέντε τρεις τρίτες χώρες, δηλαδή την Αυστραλία, τον Μπρουνέι, την τον Καναδά, την Ιαπωνία και τις Ηνωμένε Πολιτείε. Από τον Απρίλιο λοιπόν του 2014 ξεκίνησε αυτή η περίοδος των έξι μηνών και εγκρίθηκε μια πρώτη έκθεση τον Οκτώβριο του 2014 και ανάμεσα στον Απρίλιο και τον Οκτώβριο του 2014 δημιουργήσαμε ένα πλαίσιο τριμερών επαφών όπου λάμβαναν μέρος τα πέντε αυτά κράτη-μέλη και οι πέντε τρίτες χώρες και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προσπαθούσαμε να καταλήξουμε σε κάποια μέτρα προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση, να γίνει μια ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά τις πολιτικές θεωρήσεων που ακολουθούν από τη μια τα κράτη-μέλη και από την άλλη οι τρίτες χώρες και να δούμε τελικά θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε μια επίσημη απόφαση για την ελευθέρωση των θεωρήσεων. Τον Οκτώβριο λοιπόν 2014 εγκρίθηκε η πρώτη επίσημη έκθεση και στη συνέχεια εγκρίθηκε και μια δεύτερη έκθεση τον Απρίλιο του 2014. Κανένα από τα κράτη-μέλη βέβαια της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ζήτησε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναστείλει το καθεστώς ε, μη υποχρέωσης θεώρησης για αυτές τις ε, πέντε τρίτες χώρες. Πλησιάζει η επόμενη προθεσμία, θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς έχουν τώρα τα πράγματα και τι θα γίνει όσον αφορά τις υφιστάμενες περιπτώσεις μη αμοιβαιότητος. Τα θετικά νέα είναι ότι αυτές οι περιπτώσεις μη αμοιβαιότητος με τον Μπρουνέντα Ρουσαλάμ έχουν επιληθεί. Ωστόσο, τα αρνητικά νέα είναι ότι όσον αφορά τον Καναδά ιδίω και όσον αφορά τις Ηνωμένε Πολιτείες Αμερικής, εκκρεμούν ακόμα οι περιπτώσεις αυτές μη αμοιβαιότητος όσον αφορά την πολιτική θεωρήσεων και για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, δεν νομίζω ότι πρόκειται να επιληθούν οι περιπτώσεις αυτές πριν τον Απρίλιο του 2016, όταν δηλαδή θα χρειαστεί να εγκρίνουμε μια κατεξοδότηση πράξη. Όσον αφορά τις Ηνωμένε Πολιτείε, ξέρετε ότι στα πλαίσια της εσωτερικής νομοθεσίας τους προβλέπουν συγκεκριμένες νομικές προϋποθέσεις όσον αφορά το πρόγραμμα Visa Waiver, δηλαδή το καθεστώς απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης. Υπάρχει υψηλό ποσοστό απόρριψης θεωρήσεων, το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο 3% και τα δύο, ή μάλλον τα πέντε κράτη-μέλη που επηρεάζονται, Βουλγαρία, Ρουμανία, Κύπρος, Κορατία και Πολωνία, είναι χώρες ε, οι οποίες απέχουν από το κατόφλι αυτό και δεν νομίζω ότι θα καταφέρουν να περάσουν ή να ε, κατεβούν κάτω από το κατόφλι αυτό πριν τον Απρίλιο του 2016. Ανάλογη είναι και η κατάσταση στον Καναδά, δηλαδή οι ε, Καναδοί μόλον ότι δεν είναι τόσο αυστηροί στη δική τους εσωτερική νομοθεσία και αυτοί χρησιμοποιούν μια σειρά από κριτήρια και πιο συγκεκριμένα τα κριτήριά τους είναι ποσοτικά και ένα από τα κριτήρια είναι το ποσοστό απόρριψης θεωρήσεων και ένα άλλο κριτήριο είναι καταχρηστική μετανάστευση. Προσπαθούν να υπολογίσουν λοιπόν ένα μέσο όρο για τους δείκτες αυτές σε τριετή περίοδο και τα κράτη-μέλη τα οποία Ρουμανία και Βουλγαρία δηλαδή, τα οποία πρέπει να έχουν θεωρήσεις για τον Καναδά, θα πρέπει για μία τριετή περίοδο να βρίσκονται κάτω από το κατόφλι στα κριτήρια αυτά που έχουν θέσει ο Καναδάς και οι Ηνωμένε Πολιτείε. Για άλλη μια φορά λοιπόν και για τον Καναδά δεν νομίζουμε ότι πριν τον Απρίλιο 2016 θα καταφέρουν οι χώρες αυτές να βρεθούν κάτω από το κατόφλι αυτό. Έτσι έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Όπως σας είπα λοιπόν, κατά πάσα πιθανότητα τον Απρίλιο 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα χρειαστεί να εγκρίνει μία κατεξοδότηση πράξη μέσω της οποίας θα επιβάλλει υποχρέωση θεώρησης για τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα ήθελα επίσης ε, να επιστήσω την προσοχή σας ε, σε ένα πιο συγκεκριμένο τώρα σημείο και σας ενθαρρύνω πραγματικά να διαβάσετε τις δύο εκθέσεις που έχουμε ήδη υιοθετήσει, όπου σε εξηγούμε κάθε δυνατή λεπτομέρεια την κατάσταση. Θα ήθελα να αφαιρθώ λοιπόν στην περίπτωση των απαιτήσεων θεωρήσεων που έχει επιβάλει τώρα η Ιαπωνία στους κατόχους προσωρινών διαβατηρίων από τη Ρουμανία. Το ζήτημα το οποίο τίθεται και το θέσαμε και στις δύο εκθέσεις στις οποίες αναφέρθηκα, δεν ξέρουμε λοιπόν αν αυτό εμπίπτει πραγματικά στο πεδίο εφαρμογής του αναθεωρημένου μηχανισμού μία αμοιβαιότητος. Το συζητήσαμε με τα κράτη-μέλη στα πλαίσια των συζητήσεων αυτών που είχαμε στο Συμβούλιο. Δεδομένου όμως ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι συνομοθέτης, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίσουμε και ποια είναι η άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προτού λάβει οποιαδήποτε οριστική απόφαση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για το αν δηλαδή το ζήτημα αυτό εμπίπτει στο μηχανισμό αμοιβαιότητος. Δεν θα ήθελα τώρα να σε εξηγήσω για ποιο λόγο κλείνει υπέρ τη μία ή τη άλλη απόφαση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν έχουμε χρόνο άλλωστε για να κάνουμε κάτι τέτοιο. Ήθελα απλώ να επιστήσω την προσοχή σα στο ιδιαίτερο αυτό ζήτημα και θα ήθελα να ακούσω και την άποψη των συναδέλφων σα. Ευχαριστώ πολύ. Okay, thank you very much. Um, Ευχαριστούμε πολύ. Ε, που έγιναν ε, καθυστερήσεις. Ε, να ζητήσω λοιπόν από τα μέλη να μου κάνουν ερωτήσεις αν υπάρχουν προς την Επιτροπή. Όχι. Τους αφήνουμε έτσι πολύ ελαφρά σήμερα να την περάσουν. Ωραία. Υπάρχει κάποιος άλλος από την Επιτροπή που θέλει να μιλήσει. Θέλατε να μιλήσετε και οι δύο σας. Για, την, για το Περού και την Κολομβία. Ναι, αν συμφωνείτε και πρόεδρε να σας δώσω μια σύντομη παρουσίαση για τη Γεωργία και την Ουκρανία και μετά για την κατάσταση μετά την απελευθέρωση των θεωρήσεων στα Δυτικά Βαλκάνια. Για την Γεωργία και την... να γνωρίζετε ότι ο διάλογος ξεκίνησε το 2012 με ένα σχέδιο δράσης για την απελευθέρωση των θεωρήσεων των Φεβρουάριο του 2013 συμφωνήθηκε αυτό. Η Γεωργία εργάζεται από αυτού έκτοτε και με την παρακολούθηση και υποστήριξη της Επιτροπής. Η τελευταία έκθεση, η δεύτερη έκθεση πρόοδου εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2014 και πραγματικά το συμπέρασμα ήταν ότι η Γεωργία είχε κάνει τις απαραίτητες νομικές ε, αλλαγές, μεταρρυθμίσεις και στο ε, πεδίο πολιτικής μπορούσαμε να προχωρήσουμε παραπέρα και να πάμε στη φάση της εφαρμογής. Ε, επίσης, στις 8 Μαΐου εγκρίθηκε η έκθεση όπου ε, γινόταν αξιολόγηση των διαφόρων ε, σημείων στοιχείο είναι για την γεωργία σχετικά με την εφαρμογή και είχαμε και συνεργασία με τους εμπειρογνώμονες για το θέμα αυτό. Στο συμπέρασμα της η έκθεση λέει ότι η πρόοδος της γεωργίας ήταν όντως ε, σημαντική. Υπάρχει μεγάλη δέσμευση από την πλευρά της γεωργίας να υπάρξει πρόοδος ε, σε όλα τα επίπεδα των συγκρίσιμων κριτηρίων, των benchmarks ε, γενικά θεωρείται ότι έχουν επιτευχθεί τα περισσότερα benchmarks. Ε, ένας μεγάλος αριθμός επίσης έχει σχεδόν επιτευχθεί. Υπάρχουν κάποια που είναι, ε, η επίτευξη έχει γίνει εν μέρη. Ας πούμε το άσυλο, το εμπόριο ανθρωπίνων όντων, ναρκωτικών και η πάταξη της διαφθοράς. Λέει η έκθεση λοιπόν ότι θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε και να παρακολουθούμε τη γεωργία σε αυτή τη διαδικασία και η επόμενη έκθεση θα εκδοθεί στα τέλη αυτού του έτους. Αυτό σημαίνει ότι μέσα στο καλοκαίρι έγινε μια σειρά συναντήσεων με τις αρχές της γεωργίας για την υποστήριξή τους όσον αφορά στην εφαρμογή των εκκρεμών στοιχείων και συστάσεων. Πήραμε ενημέρωση από τη Γεωργία σχετικά με το πού βρίσκονται και υπήρξαν και κάποιες αποστολές οι οποίε θα γίνουν περίπου στο τέλος αυτών των μήνα για να δούνε τι γίνεται στο πεδίο, οπότε μέχρι τα τέλη του έτους θα μπορέσουμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται με τα benchmarks που εκκρεμούν. Τώρα για την Ουκρανία. Ο διάλογος ξεκίνησε το 2008 με το σχέδιο δράσης να συμφωνεί το 2010. Η Ουκρανία είναι στη δεύτερη φάση και αυτή της απελευθέρωσης των θεωρήσεων την ίδια μέρα, λοιπόν, εγκρίναμε την πέμπτη έκθεση προόδου, δηλαδή στις 8 Μαΐου του 2015. Συνολικά, η Ουκρανία φαίνεται ότι έχει κάνει εξουσιομοίωτη πρόοδο, ειδικότερα λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρετικές συνθήκες και τις εσωτερικές και εξωτερικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα Εν τούτης υπάρχει μια σειρά πεδίων ε, στα οποία η Ουκρανία ενθαρρύνεται να συνεχίσει τις προσπάθειές της ε, και να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις. Μεταξύ αυτών υπάρχουν διάφορα benchmarks που έχουν είτε εν μέρη επιτευχθεί είτε σχεδόν επιτευχθεί Θεωρούμε ότι αυτό δίνει καλές προοπτικές για την περαιτέρω πρόεδρο. Για ε, αυτά που έχουν μέρη επιτευχθεί είναι η μετανάστευση, το άσυλο, η πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος, ε, το εμπόριο ανθρωπίνων όντων και η πάταξη της διαφοράς ε, όπως και το εμπόριο των ναρκωτικών. Όσον αφορά στη διαδικασία έχουμε την ίδια με αυτή της Γεωργίας. Είχαμε στενές επαφές το καλοκαίρι. Ξεκίνησαν αυτή την εβδομάδα οι αποστολέ αξιολόγηση. Θα συνεχίσουμε το Σεπτέμβρη και περιμένουμε η επόμενη έκθεση προόδου να εκδοθεί μαζί με αυτή τη γεωργία, δηλαδή πριν το τέλος του έτους. Ε, θα δείχνει λοιπόν πώς έχουν τα πράγματα στο πεδίο ε, σε εκείνη τη φάση. Το τελευταίο που θα ήθελα να θίξω εγώ είναι η πέμπτη έκθεση για την κατάσταση σχετικά με την κατάσταση μετά την απελευθέρωση των θεωρήσεων στα Δυτικά Βαλκάνια. Υπάρχουν δύο φάσεις, το 2009 και το 2010. Βάσει αυτών των φάσεων έγινε άρση της, ε, των θεωρήσεων σε όλα τα Δυτικά Βαλκάνια εκτός από το Κωσυφοπαίδιο. Η Κομισιόν έκτοτε, παρακολουθεί έκτοτε την κατάσταση σε στενή συνεργασία με την ΕΑΖΟ και τη Frontex. Κάποια γενικά σχόλια σχετικά με αυτό. Καταρχάς πρέπει να τονίσουμε ότι η επίπτωση της απελευθέρωσης ήταν πολύ θετική. Ενθαρρύνθηκαν ε, ε, ε, τα καλόπιστα ταξίδια και γενικά οι μετακινήσεις προς την Ευρώπη. Θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω για το νούμερο του 2015 και να μην μείνω τα νούμερα που υπάρχουν στην έκθεση, γιατί αυτός ο στόχος είναι, κινείται πολύ γρήγορα. Ε, καταρχάς αυτή η έκθεση καλύπτει την κατάσταση όσον αφορά τους ε, ε πολίτες των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Δεν μιλάμε για τις ροές προσφύγων όπως είναι οι Σύριοι που ε, περνάνε από εκεί για να φτάσουν στην Ευρώπη. Δεν είναι θέμα σε αυτή την έκθεση. Όσον αφορά στα Δυτικά Βαλκάνια λοιπόν και τους πολίτες αυτών των χωρών θα ήταν χρήσιμο να δούμε λίγο τις αναλογίες. Ε, γιατί ε, όταν το συγκρίνουμε αυτό με τις μεγαλύτερες κρίσεις που έχουμε για άλλες εθνικότητες και σε σχέση με τους Σύριους θα πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη. Έτσι λοιπόν το 2014 ήταν άλλο ένα έτος αύξησης όσον αφορά στην αιτήσει ασύλου. Είχαμε 70.000 αιτήσει στα Δυτικά Βαλκάνια συνολικά. Τα βασικά κράτη-μέλη στα οποία κατατέθηκαν για τα οποία κατατέθηκαν αιτήσει ήταν η Γερμανία, η Σουηδία, η Γαλλία και το Βέλγιο. Αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Το 2015 φαίνεται ότι τα νούμερα θα συνεχίσουν να αυξάνονται. Στους πρώτους πέντε μήνες είχαμε ήδη 33.000 αιτήσει, δηλαδή σε σχέση με το 2014, την ίδια περίοδο, έχουμε διπλάσεις και παραπάνω αιτήσει. Φέτος λοιπόν η τάση δείχνει ότι οι Αλβανοί είναι αυτοί που ε, απαριθμούν τα περισσότερα μέλη σε σχέση με άλλες ε, εθνικότητες. Ε, πέρυσι ε, ήταν οι Σέρβοι, φέτος οι Αλβανοί είναι η πλειονότητα. Όσον αφορά τα ποσοστά αναγνώρισης στα κράτη-μέλη, είναι πολύ χαμηλά, δηλαδή ε, μικρό ποσοστό για όλες τις εθνικότητες είναι λοιπόν μια σημαντική τάση που συνεχίζουμε να παρακολουθούμε στενά. Η έκθεση κάνει μια σειρά συστάσεων σχετικά με το πώς να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα που παραμένουν ε, ακόμα ενισχύ. όσον αφορά τα Δυτικά Βαλκάνια ενθαρρύνονται για να έχουν ένα σύστημα το οποίο θα βοηθά στην επιχειρησιακή συνεργασία με τα κράτη-μέλη, θα καταγράφει καλύτερα τα διάφορους ετούντες άσυλο, θα ε, μπορεί να αντιμετωπίζει την παράνομη διακίνηση μεταναστών, θα προωθεί την σεβασμό των θεμελιωδών ε, δικαιωμάτων και θα κάνει και στοχευμένες εκστρατείες σχετικά με τα δικαιώματα που έχει ο κάθε άνθρωπος που θέλει να ταξιδέψει στην Ευρώπη. Επίσης υπάρχουν συστάσεις τα κράτη-μέλη που έχουν τις περισσότερες αιτήσει σχετικά με την εξορθολογισμό των διαδικασιών για το άσυλο, αλλά και εξαρτής πληροφόρηση σε αυτές τις χώρες επίσης. Το επόμενο βήμα που παρασκευάζεται αυτή τη στιγμή είναι ε, μια λίστα ασφαλών χωρών προέλευσης που περιλαμβάνει και τις χώρες των Βαλκανίων. Θα σταματήσω λοιπόν εδώ και είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Μία άμεση ερώτηση είναι οι αιτήσει ασύλου που αυξάνονται θα έχει επίπτωση στην αφιλελευθερωπήση θεωρήσεων διαβατηρίων για τα Δυτικά Βαλκάνια. Αυτή είναι μια ερώτηση που θα ήθελα να διατυπώσω. Συνάδελφοι, αν έχετε ερωτήσει προ την Επιτροπή, τώρα είναι η ώρα για κάποιο από τα συγκεκριμένα αυτά τα θέματα. Για το Περού και την Κολομβία που τον Ιούνιο είχαμε το αρχικό στάδιο. Πρέπει να γνωρίζουμε πώς έχει εξελιχθεί η κατάσταση πρωτού προχωρήσουμε. Για άλλα θέματα κάποιος που θα ήθελε να παρέμβει. Αν δεν υπάρχει κανείς. Θα θέλατε να επεκταθείτε και να μας επεξηγήσετε σε σχέση με τις επιπτώσεις ε, της αύξησης του αριθμού ετούντων άσυλο για τι θεωρη, ε, τις θεωρήσεις διαβατηρίων στα Δυτικά Βαλκάνια. Ναι, ευχαριστώ. Να πω ότι συνεχίζονται οι συζητήσει με τα κράτη-μέλη που βρίσκονται υπό εξέλιξη με τα κράτη-μέλη. Υπάρχει ένα μηχανισμό, όπω γνωρίζετε, όπου μπορούν να αναγνωστοποιούν ε, τα κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα θέματα για να ξεκινήσει η λειτουργία αυτού του μηχανισμού Αυτά σε σχέση με τον αγωνισμό που βρισκόμαστε. Συνεχίζουμε την του συζήτηση με τα κράτη-μέλη. Έχουμε συναντήσεις και θα έχουμε συναντήσεις και με τα κράτη των Δυτικών Βαλκανίων. Αυτή είναι η κατάσταση που έχει τώρα σχετικά. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε πολύ για τόσα όσα μας είπατε. Ευχαριστούμε λοιπόν. Περού Κολομβία τώρα. Μπορείτε σύντομα να μας τα αναφέρετε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τώρα για μένα είναι αυτό το θέμα. Όπως γνωρίζετε έχουμε τον κανονισμό 539 του, που τροποποιήθηκε το Μάιο 2014 και η μεταφορά στον θετικό πίνακα κρατών που συμπεριλάμβανε ιδιαίτερα ε, μια, μικρά κράτη στην Καραϊβική και στον ε, Ειρηνικό καθώς επίσης ε, και τα Αραβικά Εμμυράτα, το Περού και την Κολομβία. Από τους συνομοθέτες εγκρίθηκε το Μάιο 2014 και φυσικά η υποαίρεση ότι αυτό το θέμα θα συμπεριληφθεί σε σχέση με την άρση απέτησης χορήγησης θεωρήσεων διαβατηρίων για αυτές τις χώρες. Η Επιτροπή είχε κατευθυντηρίες γραμμές για τις διαπραγματεύσεις το Περού και η Κολομβία έχουν μια διαφορετική ιστορία ωστόσο όμως ε, για τα υπόλοιπα έχει οδηγίες από το Συμβούλιο η Επιτροπή για την έναρξη διαπραγματεύσεων για την απαλλαγή θεωρήσεων διαβατηρίων για αυτές τις χώρες από το φθινόπωρο δηλαδή 2014 πέρυσι ήδη και πολλές από αυτές τις διαπραγματεύσεις ε, στέφθηκαν με επιτυχία και ολοκληρώθηκαν γοργά και μια επιστολή σχετικά πεστάλη προς τον πρόεδρο της δικής σας κοινοβουλευτικής επιτροπής από τον δικό μου γενικό διευθυντή στις 27 Μαρτίου 2015. Και τώρα βλέποντας ότι οι διαπραγματεύσεις ε, που όπως το ανέφερα για τα πρακτικά με την Δομινίκη, Γρανάδα, Αγία Λουκία, Άγιο Βικένδιο, Τιμό Λέστε, Τρινιδάτ και τον Πάγκο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Βανουάτου, ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν και έχουν μονογραφεί συμφωνίες και προβλέπονται προσωρινά, προσωρινά οι αιτήσει εφαρμογής αυτών των διατάξεων μέχρι την τελική μερομηνία κύρωσης και σε σχέση με την επιστολή που ενημέρωνε για το πώς είχαν οι διαπραγματεύσεις όλες αυτές οι διαπραγματεύσεις πράγματι μεταξύ έχουν υπογραφεί και έχουν αρχίσει να ισχύουν φυσικά με αναμένοντας την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες όπως το επιπέρου και Κολομβία κάπως διαφορετική κατηγορία τους. Την τελευταία στιγμή προσθέθηκαν στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υποπίεση αρκετών κρατών μελών και άλλων εμπλεκομένων μελών η συμπερίληψη του Περού και της Κολομβίας σε αυτή την τροποποίηση ήταν υπό την αίρεση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρώτα θα διεξήγαγε μια αξιολόγηση του πώς έχουν ε, προχωρήσει τα πράγματα για να δικαιούνται την απαλλαγή θεωρήσεων διαβατηρίων αυτές οι χώρες. Δηλαδή πρέπει να αξιολογήσει ακόμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα κριτήρια τα οποία συμπεριλαμβάνονται για τις διατάξεις ε, για την απαλλαγή χορήγησης ε, θεωρήσεων διαβατηρίων. Οι εκθέσεις ε, τον Οκτώβριο πέρυσι ε, ολοκληρώθηκαν και συνήγαγε το συμπέρασμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι παρότι υπήρχαν προβλήματα ακόμα με τα ναρκωτικά και το οργανωμένο έγκλημα, συνολικά θεωρήθηκε ότι αυτές οι χώρες θα μπορούσαν να εξεταστούν ως επιλέξιμες για την απαλλαγή θεωρήσεων διαβατηρίων. Στη συνέχεια η διεξαγωγή διαπραγματεύσεων συνεχίστηκε με αυτές τις χώρες και το, την άνοιξη εφέτος διαπραγματευτήκαμε, συνεχίσαμε τις διαπραγματεύσεις μαζί τους που αρχικά αυτές οι δύο ε, συμφωνίες στο περιθώριο της ε, Συνόδου ε, Κορυφής στις Βρυξέλλες μπόρεσαν να εξεταστούν και να προχωρήσουν. Για το Περού και την Κολομβία προσβλέπουμε τώρα στην επίσημη υπογραφή της συμφωνίας. Την επόμενη εβδομάδα θα εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το σχέδιο αποφάσεων του Συμβουλίου για την ολοκλήρωση αυτών των διατάξεων απαλλαγής χορηγήσεων θεωρήσεων διαβατηρίων καθώς και για τα άλλα νησιά και είναι πια στα χέρια του Συμβουλίου να εγκρίνει το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου και αυτές οι δύο συμφωνίες θα αρχίσουν να ισχύουν από την ημερομηνία υπογραφής αυτών των πράξεων οι συμφωνίε θα αρχίσουν να ισχύουν. Αυτά σε σχέση με τι διεθνεί ε, συμφωνίε και διαπραγματεύσει Με ικανοποίηση πρόθυμο σήμερα να δώσω περισσότερε λεπτομέρειε αν κάποια μέλη το επιθυμούν. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σα ευχαριστώ. Χουαν Φερνάντο, εσύ θα ήθελε να αναφέρει κάτι. Παρακαλώ. Χουαν Φερνάντο Λόπεθ Αγιλάρ. Ναι, Πρόεδρε, για αυτό το σημείο ιδιαίτερα, αν μου επιτρέπετε να λάβω τον λόγο για το Περού και την Κολομβία, για να δώσω κάποια συνέχεια σε αυτό το θέμα, διότι μάλιστα κάποια μέλη της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών της ΛΥΜΕ είχαν δραστηριοποιηθεί ιδιαίτερα όταν υπήρξε η καθυστέρηση ε, στα χαρτοφυλάκια Περού και Κολομβίας για την διαδικασία απελευθέρωσης από τις ε, χορηγήσεις δια, ε, θεωρήσεων διαβατηρίων. Από τότε όμως δεν ενημερωθήκαμε, δεν έχουμε κάποιες πληροφορίες στα χέρια μας. Και σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 10 για την περίπτωση Μαυρικίου, Μωρίσιος... είναι σαφές ότι το Ευρωκοινοβούλιο έχει δικαίωμα να ενημερώνεται με ακριβείς πληροφορίες σε τακτά διαστήματα και όχι μόνο μετά από αίτημα δικό του, αλλά και με πρωτοβουλία των ιδίων θεσμικών οργάνων αυτοβούλος, αυτοδικαίως. Θα ήθελα εδώ να προσθέσω το ότι όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα θα πρέπει τουλάχιστον να δούμε πώς έχει το χρονοδιάγραμμα ένταξη σε ισχύ αυτής της πολιτικής απόφασης που ελήφθη και ενεκρίθη από την Επιτροπή Λίβε Πολιτικών Ελευθεριών και όσον αφορά τα θέματα εξωτερικής πολιτικής αυτές οι χώρες, για αυτές τις χώρες Κολομβία και Περού και για τις επιπτώσεις που υπάρχουν και για κάποιες άλλες χώρες που θα μπορούσαν να, να αιτηθούν το ίδιο καθεστώς αλλά τουλάχιστον για την Κολομβία και το Περού να γνωρίσουμε ποιο είναι το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. Γνωρίζουμε ότι και οι δύο συμφωνίες επικυρώθηκαν κατά το πρόσφατο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Συνόδου Κορυφής του Ιουνίου μεταξύ ΕΕ και κρατών της Λατινικής Αμερικής. Όμως έκτοτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ενημέρωσε το Κοινοβούλιο σχετικά και ούτε είχαν παρασχεθεί αυτές οι πληροφορίες προηγούμενα, ούτε πριν ούτε μετά. Έτσι λοιπόν το ζήτημα είναι ότι θα επιθυμούσαμε εμείς να, πώς να το πω, να ενημερωθούμε, να γνωρίζουμε πώς έχει εξελιχθεί, πώς έχουν τα πράγματα τώρα και να έχουμε μια σαφή εικόνα τι ακριβώς συμβαίνει με το χρονοδιάγραμμα για κάθε έναξη ε, σε ισχύ αυτών των συμφωνιών επιμέρους Αναφέρατε κάπως και είπατε τα διαδικαστικά βήματα τα οποία θα πρέπει να ακολουθηθούν. Αλλά δεν υπάρχει σαφής εικόνα για το χρονοδιάγραμμα. Ποιο θα ήταν αυτό το χρονοδιάγραμμα. Το προβλεπόμενο, εκτιμόμενο αυτό χρονοδιάγραμμα. Και με την καθυστέρηση που θα συνεπάγεται για την έναξη σε ισχύ τελικά μετά από όλα αυτά αυτή της συμφωνίας. Ευχαριστώ. I think, ε, λοιπόν, Νομίζω ότι οι απαντήσεις στις ερωτήσεις σας εξαρτώνται περισσότερο από το Συμβούλιο και όχι τόσο πολύ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ας ακούσουμε όμως και την παρατήρηση της Μαρή Κριστίν και μετά θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μαρή Κριστίν, έχει το λόγο. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε σημαντικές τακτικές επαφές για το ζήτημα αυτό. Ήδη τον Ιούλιο μας είχε γίνει μια πρώτη ενημέρωση Μα είχε παρουσιαστεί τότε μια έκθεση που ήταν ακόμα σε εξέλιξη και τότε, αν θυμάστε τον Ιούλιο, πολλοί συνάδελφοι είχαμε πει ότι λυπούμασταν πάρα πολύ, πάρα πολύ που βρισκόμασταν μπροστά από ένα τετελεσμένο γεγονό. γιατί ήδη είχε εγκριθεί τότε συμφωνία χωρί να έχει δώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη δική του τη γνώμη. Τώρα μιλάμε για το Περού και για την Κολομβία και γενικότερα έχω την εντύπωση ότι ήμασταν υπέρ της ελευθέρωση των θεωρήσεων προς συγκεκριμένους τουριστικούς προορισμούς και ότι προσπαθούσαμε ουσιαστικά να προωθήσουμε τα συμφέροντα των Ευρωπαίων τουριστών. Τώρα έχουμε τα Ενωμένα Αραβικά Εμμυράτα, πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί, και τώρα ξαφνικά σε αυτόν τον κατάλογο βλέπω και το Περού και την Κολομβία. Αφενό με, λοιπόν θέλω και εγώ να γνωρίζω ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα, βρισκόμαστε σε απόφαση. Αυτό θα έλεγα ότι είναι προσβλητικό απέντη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και αν κατάλαβα καλά, ουσιαστικά ήταν ε, η σύνοδος ΣΕΛΑΚ με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής που υποκίνησε την όλη αυτή προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τι υπόθηκε εκεί, τι έγινε εκεί και κινητοποιήθηκε τόσο πολύ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τι μέτρα έχετε λάβει προκειμένου να καταστήλετε το εμπόριο ναρκωτικών, το οποίο όπως ξέρετε ε, είναι έντονο φαινόμενο σε αυτές τις δύο χώρες. Τι έχει γίνει έκτοτε λοιπόν. Σε ευχαριστούμε Μαρία Κριστίνα. Να ξαναδώσω τώρα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να πω και εγώ με τη σειρά μου ότι όντως ε, θελήσαμε κι εμείς να έχουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων διότι έχουμε και εμείς συγκεκριμένε ανησυχίες επί της διαδικασίας, αλλά και επειδή σύμφωνα με το άρθρο 218 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ενημερώνεται σε τακτική βάση και επισήμως για όλες αυτές τις ανεξελίξει διαπραγματεύσεις για τις συμφωνίες. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο θέλησαν να έχουμε σήμερα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί μα και στο μέλλον θα είναι πολύ σημαντικό να συνεχιστεί και αυτή τη διαδικασία. Να είναι δηλαδή υπόλογη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τι αποφάσει αυτέ. Ενδεχομένω οι δύο εκπρόσωποι τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελαν να απαντήσουν στου δύο συναδέλφου. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα για τη θέση σε ισχύ των συμφωνιών απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρηση για την Κολομβία και το Περού. Όπω σα είπε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εγκρίνει ένα σχέδιο απόφαση στι 14 Σεπτεμβρίου. Στη συνέχεια η απόφαση αυτή θα διαβιβαστεί στο Συμβούλιο και εκεί βέβαια θα πρέπει να εγκριθεί από τα κράτη-μέλη αυτή η απόφαση. Αυτή τη στιγμή οι περισσότερε χώρε αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν ήδη πει ότι είναι υπέρ τη ελευθέρωση θεωρήσεων για τι δύο αυτέ χώρε θεωρούμε ότι θα είναι μια τυπικότητα η έγκριση από το Συμβούλιο. Νομίζω λοιπόν ότι κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου θα πρέπει να καταφέρουμε να βρούμε μία ημερομηνία με τις δύο αυτές χώρες προκειμένου να υπογραφεί επισήμως συμφωνία, γιατί ξέρετε ότι απλώς ξεκίνησε η όλη διαδικασία στην σύνοδο EU-SELAC. Ουσιαστικά οι επικεφαλείς διαπραγματευτές συμφώνησαν επί της αρχής για το κείμενο, πρέπει πάντως να υπογράψουν επισήμως και δύο χώρες μέχρι το τέλος του 2015 και θα εφαρμόζονται οι αποφάσεις αυτές προσωρινά μέχρι να τεθούν επισήμως σε ισχύ αυτή τη στιγμή σε εγκριθεί επισήμως και συμφωνία. Αυτά όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα. Ο γενικός μου διευθυντής ξέρω ότι έχει έρθει τον Νοέμβριο στη δική σας την Επιτροπή και μεταξύ άλλων σας ενημέρωσε για το Περού και για την Κολομβία όσον αφορά τις εκθέσεις αξιολόγησης που είχε τότε εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επίσης ενημέρωσε την Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την πρόοδο που είχε σημειωθεί μέχρι τότε για το ζήτημα της ελευθέρωσης των θεωρήσεων. Επίσης μια επιστολή απεστάλλει ήδη την Άνοιξη του 2015 στην Επιτροπή σας. Νομίζω εν γέννη ότι η Επιτροπή σας έχει ενημερωθεί καταλήλως, πλήρως και συστηματική βάση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή εμπλέκεται στη διαπραγματεύση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξυπακούεται ότι θα πρέπει να ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδίω τη δική σα την Επιτροπή τόσο για την έκβαση των διαπραγματεύσεων, όσο και για προβλήματα που ενδεχομένω να προκύπτουν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Για αυτό το λόγο λοιπόν βρίσκομαι εδώ σήμερα, αλλά και ο γενικός μου διευθυντής, όπως σας είπα, μέσω μίας επιστολής στην Άνοιξη, σας ενημέρωσε για τα όσα λέμε σήμερα. Τι συμβαίνει δηλαδή με το Περού και την Κολομβία, σε ποιο στάδιο διαπραγματεύσεων βρισκόμαστε. Ολοκληρώνοντας να σας πω ότι ε, εμείς ε, είμαστε στη διάθεσή σας ανα πάσα στιγμή να ερχόμαστε εδώ πέρα και να σας ενημερώνουμε για οποιοδήποτε ζήτημα σας απασχολεί στα πλαίσια της πολιτικής θεωρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταλαβαίνω ότι στη δική σας την Επιτροπή πρέπει να εξετάζονται αυτά τα ζητήματα. Είμαστε λοιπόν στη διάθεσή σας για να σας δώσουμε περαιτέρω λεπτομερείς πληροφορίες ανα πάσα στιγμή. Ευχαριστώ πολύ. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τους συναδέλφους που πήραν το λόγο. Νομίζω ότι εδώ ε, φτάσαμε στο τέλος αυτής της συζήτησης. Ευχαριστούμε και ε, όλους εσάς ε, που ήσασταν εδώ σήμερα, γιατί εδώ τελειώνει η ημερήσια διάταξη. Υπάρχουν στα λοιπά κάποια θέματα. Στις 30 Σεπτεμβρίου στις 14 και 15 Σεπτεμβρίου, συγγνώμη, έχουμε τις επόμενες συνεδριάσει. Ε, τελειώσαμε λίγο νωρίς σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ σε ευχαριστώ.